Ξεκινάμε την συνεδρίαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ωραία. Θα ήθελα να συμπληρώσω πως ε, είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε γιατί υπήρχαν ε, φήμες πως ε, ο Επίτροπος Σεύκοβιτς τον οποίον εγκρίναμε ομοφόνος, ε, ίσως καταλήξει κάπου αλλού και να είναι άλλος ο αρμόδιος επίτροπος. Γι' αυτό μίλησα με όλους τους ε, συντονιστές ε, και είπαμε να γράψουμε μια επιστολή στον Γιούνκερ και να πούμε πως εμείς θέλουμε να διατηρήσει αυτή την θέση και να μην αλλάξει χαρτοφυλάκιο για να μην χρειαστεί, και να μην χρειαστεί να κάνουμε και άλλη ακρόαση. Και οι 7 συντονιστές ε, συμφώνησαν. Ε, έστειλα την επιστολή και στον Γιούνκερ και στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να έχουμε θετική αντίδραση και να μην αλλάξει τίποτα. Το έστειλα σε όλους τους ε, συντονιστές και αν θέλετε να το διαβάσετε, ρωτήστε, ζητήστε παρακαλώ την επιστολή από τους συντονιστές σας δόθηκε και στον τύπο και Ελπίζω πράγματι να μην ε, χρειαστεί να κάνουμε καινούργια κρόαση. Ωραία, λοιπόν. Τα πρακτικά της 3ης Σεπτεμβρίου, εάν δεν υπάρχει ε, καμία αντίρρηση, επίσης εγκρίνονται. Οι αποφάσεις ε, των συντονιστών από τις 3 και 18 Σεπτεμβρίου είναι επίσης στην διάθεσή σας. Εάν μέχρι τις 6 το απόγευμα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, εγκρίνονται. Καλώς. Οπότε περνάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Έχουμε αρκετές σήμερα. Γιατί ουσιαστικά διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια δοκιμαστική. Έχετε όλη την καρτούλα σας. Καλά, τέλος θα το παραβλέψουμε, αλλά στην Ολομέλεια δεν γίνονται αυτά, μόνο στην Επιτροπή. Νομίζω λύθηκε το πρόβλημα, γιατί έχει κάνα δύο παραπάνω το ΕΛΚ Λοιπόν, να δοκιμάσουμε. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Τώρα. Άμα αλλάξετε θέση ίσως. Τώρα δουλεύει. Ωραία. 39 κάρτες λοιπόν λειτουργούν. Να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Τι. Πριν. Ε, αν είναι να ψηφίζετε προφορικά πρέπει να το λέτε πριν για να μην αλλάξετε άποψη αφού δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Λειτουργούν όλα. Ξεκινάμε. Έχουμε τη διαπραγματευτική εντολή για τα έξι κομμάτια του τέταρτου σειροδρομικού πακέτου. Υπήρχαν διάφορες φήμες πώς θα το σπάσουμε. Εμείς λέμε πώς ε, θα πάνε και τα έξι μαζί. Το αποφασίσαμε ε, τον Ιανουάριο ως Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο δεν μας ακολουθεί. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε χωριστά για κάθε εντολή και απαιτείται ε, απόλυτη πλειοψηφία για το κάθε ένα από αυτά. 25 δηλαδή υπέρ. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία για βάρη και διαστάσεις. Όχι, πρώτο σειροδρομικό πακέτο. Η πρώτη ψηφοφορία ε, είναι του κυρίου Σασόλη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι σαφές. 37 υπέρ έναντι τριών, καμία αποχή, δεκτό. Δεύτερη εντολή. Εισηγητής ο Βιμ Φαντεκάμπ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι ε, πώς ψηφίζετε. Ωραία, πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. Το τρίτο μετά είναι... Ε, η κυρία Μπιλμπάου είναι η συγγήτρια. Δεν τη βλέπω. Α, εκεί μάλιστα, ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και 38 έναντι 2. Φοβερές αλλαγές. Επόμενη έκθεση. Εισηγητής ο Μιχαήλ Κράμερ, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38 έναντι 2. Καμία αποχή. Έκθεση Τσίλε. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 37, έναντι 2 και μία εποχή. επόμενη έκθεση. Έκθεση Κιλόνεν. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 36 έναντι 3 και άλλη μία 37. Ωραία. Επόμενη ψηφοφορία, οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις. Γιώργ Φρυντινό εισηγητής είναι εδώ. Όχι, αλλά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38, 39 δηλαδή, έναντι 2. Μετά, στατιστικά στοιχεία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Έκθεση Κράμερ. Άρχεται... Η με συγχωρείτε ο κύριος Κράμερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν κατάλαβα. Πέρας. 39-40 δηλαδή και μία ψήφος κατά. Επόμενη στατιστικά αγαθών που μεταφέρονται με, ε, σε πλεύσιμους ποταμούς. Βασάικ Χάουτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 39. Μια αποχή. 40 δηλαδή. Ε, με μια αποχή. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες. Έχουμε σήμερα εδώ πέρα εκπροσώπους της DG Move από την Κομισιόν για να μας ενημερώσει για μια πράξη κατεξιοδότηση για την οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα για το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου Οδήγησης. Να σας πω το εξής. Πρώτον, η οδηγία ITS 2010-40 της Κομισιόν είναι η νομική βάση για την πράξη κατεξιοδότηση για να καθορίσει τις ε, προδιαγραφές του ETS. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα διπλό δικαίωμα εξέτασης της πράξης αυτής ε, κατεξιοδότηση. Μπορεί δηλαδή είτε να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση. Δεύτερον, μπορεί να υποβάλει κάποια αντίρρηση, ένσταση και να ζητήσει νέα πρόταση από την Κομισιόν η οποία θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη αυτά τα οποία θέλει το Κοινοβουλίο. Εδώ πέρα όμως είμαστε στη φάση της ε, προετοιμασίας. Και όταν υποβληθεί επισήμως η πρόταση θα αρχίσει να μετράει και ο χρόνος για την προθεσία. Παρακαλώ λοιπόν τώρα την Κομισιόν να παρουσιάσει την διαδικασία και την πράξη αυτή κατά εξουσιοδότηση. Η κυρία Κοτσίνσκα λοιπόν θα τα κάνει αυτά. Έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να σας παρουσιάσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο εξουσιοδότηση πράξεως, διότι είμαστε ακόμα στην προηγούμενη διαδικασία της υιοθέτησης από πλευράς Κομισιόν, όμως εκτιμώ τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες μια ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, όπως ήδη εξήγησε ο Πρόεδρος, το πλαίσιο, η οδηγία ITS ε, ετέθη ισχύ τον Αύγουστο του 10 και θυμίζω ότι ενεκρίθη σε ένα πάρα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χάρη και την εξαιρετική, στην εξαιρετική συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Με τρεις βασικούς στόχους λοιπόν η οδηγία να επιταχύνει η συντονισμένη εφαρμογή και η χρήση των εφιών συστημάτων μεταφορών και σε συνδυασμό με άλλα συστήματα, ώστε να βελτιώνουμε την ε, διαλειτουργικότητα των συστημάτων ITS. Καθόρισε λοιπόν έξι στόχους προτεραιότητα, δράσεις μάλλον προτεραιότητα, εντός του πλαισίου των οποίων θα είχαμε κατεξουσίαν πράξη και οι πληροφορίες ε, σε πραγματικό χρόνο για τις μεταφορές είναι μία από αυτές. Εντός του πλαισίου των κατεξουσίαν πράξεων δεν θα ζητήσει η Κομισιόν να εφαρμοστούν οι υπηρεσίες αυτές, αλλά θα τεθεί ένα πλαίσιο συνθήκων και προϋποθέσεων εφόσον χρησιμοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Η εξουσιοδότηση αυτή προβλέπεται για 7 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2017, στα πλαίσια της οδηγίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι καταρχάς η οδηγία ETS ασχολείται με ένα καινούριο σχετικά πεδίο μεταξύ των, των σημείων διεπαφής μεταξύ συστημάτων μεταφορών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Η τεχνολογία κινείται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά κινούμεθα και σε καινοτόμα νομοθετικά ύδατα, διότι είναι σχετικά καινούργιο νομοθετικό μέσο και για την Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Λόγω για τον οποίο όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά για τις κατεξότησιν πράξεις αυτές, υπογραμμίσαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων, αλλά και με εκπροσώπους της Επιτροπής ΤΡΑΝ, που πρέπει να παρίστανται στις διαβουλεύσεις αυτές και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε με συναντήσεις όπως η σημερινή όπου σας ενημερώνουμε προ του διυπηρεσιακού διαλόγου διαβούλευσης εντός της Κομισιόν είμαστε ακόμα για την κατεύθυνση της πράξη αυτή, προτού δηλαδή αποσταλεί σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Σχετικά με την συγκεκριμένη εξουσιοδότηση για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις μεταφορές. Ασχολούμαστε με αυτό πάνω από ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε με τις ευρείες διαβουλεύσεις ενδιαφερομένων. Είχαμε 7 συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, με, την, με παρούσα τη γραμματεία της Επιτροπής σας. Και ήταν δύσκολο το έργο μας, διότι θα θυμάστε ότι η οδηγία είναι ευρύτατη στο πεδίο της, ε, περιγράφοντας τι πρέπει να συμπεριληφθεί στην εξιότηση αυτήν. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε ένα κοινό όραμα, ώστε οι ορισμοί για τα προβλήματα που υφίστανται να είναι κοινοί και αποδεκτοί από όλους, κράτη-μέλη και κομισιόν και κοινοβούλιο και πρέπει να καλύψουμε και όποια κενά υφίστανται, ώστε να έχουμε μία προσέγγιση που αφενός θα είχε συγκεκριμένα ωφέλη και αφετέρου δεν θα κατέληγε σε περιτο άχθος για τα κράτη-μέλη. Επίσης ενημερώσαμε την, ε, την αρχή προστασίας δεδομένων, γιατί έχει, αυτό ισχύει για όλες τις κατεξότητες πράξεις, θα πρέπει να ενέχεται η αρχή προστασίας των δεδομένων απολύτως στη δουλειά μας, αν και στη συγκεκριμένη εξοδότηση είναι απίθανο να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με προσωπικά δεδομένα, διότι εδώ μιλούμε για πληροφορίες κυκλοφορίας οχημάτων και όχι τόσο καταχώρησης ιδιωτικών οχημάτων, το οποίο θα γίνεται ε, μέσω ε, ε, συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συστημάτων sensor, Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή Τραν θα ενημερώνεται απολύτως για τη δουλειά που τρέχει και εξού και η παρουσίασή μου αυτή. Θα ήθελα όμως ε, να πάω περισσότερο στα περιεχόμενα της συμπράξεως ε, για την ε, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία. Πρέπει λοιπόν να διατηρούμε υπόψη ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των υπηρεσιών σχετικά με την παροχή τέτοιων πληροφοριών υποστηρίζονται και οθούνται από την αγορά. Αγορά η οποία στην ουσία, στην πραγματικότητα υφίσταται σε όλα τα κρατη και η ενημέρωση αυτή παρέχεται μέσω διαφόρων διόδων, καναλιών στους χρήστες. Αυτό που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι ότι μας λείπουν κάποια σημεία συνέχειας διασυνοριακής αλλά και εντός συγκεκριμένων κρατών μελών, είτε διότι δεν είναι διαλειτουργικά τα στοιχεία που έχουμε, είτε γιατί οι πληροφορίες ή ο μορφότυπος των πληροφοριών δεν είναι ίδιος σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης παρατηρούμε ότι κάποιες φορές η ποιότητα της ε, υπηρεσίας δεν είναι τόσο υψηλή, δηλαδή σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την αξιοπιστία των στοιχείων. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι η πρόσβαση, η επικαιροποίηση και η ανταλλαγή των στοιχείων επί των οποίων δομείται αυτό το σύστημα ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε αν θέλετε ένα κατάλληλο πλαίσιο ή κάποιες συνθήκες πλαίσιο ακριβέστερα ώστε να διευκολύνουμε την παροχή αξιόπιστων αλλά και ακριβέστερον ως προς το περιεχόμενο πληροφοριών σχετικά με την ενημέρωση αυτή σε πραγματικό χρόνο. Προτιμήσαμε μια απολύτως αναλογική προσέγγιση αφήνοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στα κράτη-μέλη ίσως ό,τι αφορά στην υλοποίηση και γι' αυτό στο κέντρο, στον πυρήνα της εξιότησης αυτής ήταν ένα εθνικό σημείο προσβάσεως που θα ήταν αν θέλετε ενιαία θηρίδα σχετικά με όλα τα δεδομένα κυκλοφορίας εντός ενός συγκεκριμένου δικτύου ή περιοχής περιφέρειας. Σχετικά με τις υπηρεσίες λοιπόν που ορίζονται στην εξιότηση αυτήν, οποιοδήποτε χρήστης θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια δεδομένα διατίθενται σε συγκεκριμένο ή πώς συγκεκριμένο θέμα, πώς αποθηκεύονται και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Το οποίο σημαίνει πρόσθετες πληροφορίες επανάχρησης σε σχέση με συγκεκριμένες συμβατικές ε, υποχρεώσεις. Το έγγραφο εργασίας, το οποίο είχατε και εσείς, αναφέρει στατικά δεδομένα, δυναμικά δεδομένα και δεδομένα κυκλοφοριακά. Στο παράρτημα θα δείτε κατάλογο παραδειγμάνων των, των ειδών αυτών, των τύπων αυτών δεδομένων, που θα συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία της πληροφορίας και για να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα μιλούμε για τα χαρακτηριστικά των οδών, της σήμανσης κυκλοφορίας, της ε, σύστασης συγκεκριμένων, συγκεκριμένης πορείας ή οδού προς αποφυγή κυκλοφοριακών συμφορήσεων, αλλά στον κατάλογο που συμπεριλαμβάνομαι στο παράρτημα, μάλλον ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός σε καμία περίπτωση, δηλαδή μπορούν τα κράτη-μέλη να τον συμπληρώνουν όταν χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Αυτό που ήδη ανέφερα είναι ότι το ουσιαστικότατο σημείο, μιλώντας για διαλειτουργικότητα των στοιχείων, είναι ένας τυποποιημένος μορφότυπος. Όταν μιλούμε λοιπόν για προσβασιμότητα από ενιαίο σημείο επαφής εθνικό, μιλούμε για συγκεκριμένο μορφότυπο που θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από τα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ για τα στατικά δεδομένα μιλούμε για τυποποιημένο μορφότιμο που θα εφηγραμμίζεται με τις διατάξεις οδηγίας Inspire, αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια. Δεν μιλούμε λοιπόν για νέους μορφοτύπους. Μιλούμε για μορφοτύπους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, είναι καλά, είναι διαδεδομένοι και γνωστοί στα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν δημιουργούμε μόνο συνθήκε πλαίσιο για την διαθυσιμότητα των στοιχείων, των δεδομένων, αλλά και για την επικαιροποίησή τους και το έγκαιρο της επικαιροποίησης αυτής. Οι πληροφορίες λοιπόν σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία είναι πολύ σημαντικές για την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων. Και υπάρχουν διατάξεις και σχετικά με την τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών. Κάτι άλλο που συζητήσαμε επί μακρόν με τα κράτη-μέλη ήταν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Μιλήσαμε για το ε, συνεκτικό οδικό δίκτυο και δίκτυο μεταφορικών συστημάτων των κρατών μελών ώστε να υπάρχει μια συνέπεια και μια εναρμονισμένη αν θέλετε ομοιογενής εμπειρία των οδηγών και των ατόμων που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Οι προϋποθέσεις τώρα αυτές της εξουσιοδότησης θα μπορούν να ισχύουν και για κάποια τμήματα που ονομάζονται ζώνες προτεραιότητας που θα μπορούσαν να είναι και τμήματα των αστικών οδικών δικτύων, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Εφόσον εγκριθεί η εξουσιοδότηση αυτή, αυτά θα ισχύουν για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ε, πληροφοριών για την κυκλοφορία μετά από μια μεταβατική περίοδο τριών μηνών. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα εγκριθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ιστορικές διαδικασίες της Κομισιόν σχετικά με την καθεοξουσιοδότηση σε αυτή πράξη, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στην ε, εισηγήτρια, την κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν. Είναι θετικό το ότι εμπλέκεται το Κοινοβούλιο τόσο νωρίς στην διαδικασία των πράξεων κατεξιοδότηση. Εμείς ε, θεωρούμε επί της αρχής πως αυτά τα συστήματα είναι θετικά, μπορούν να μειώσουν την κίνηση, την κατανάλωση κτλ. Έχω κάποιες ερωτήσεις τώρα. Αφενός, μιλάμε για εναρμόνιση δεδομένων και ειδικά ε, για τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται ήδη από τα κράτη-μέλη. Λογικό αυτό. Το, η ερώτησή μου είναι πόσο κοστίζει αυτό και ποιος πληρώνει. Μία ερώτηση είναι αυτή. Και κατά πόσον προκύπτουν ε, μετά δαπάνες για τον ιδιωτικό τομέα και αν μπορείτε να τις ε, ποσοτικοποιήσετε και κάτι άλλο. Όταν συλλέγονται δεδομένα, ε, τίθεται ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εγώ είμαι υπέρ της καινοτομίας και της διάθεσης των δεδομένων και της ανταλλαγής τους. Μιλήσατε και για επαναξιμοποίηση. Πράγματι πρέπει να επαναξιμοποιούνται. Το ερώτημα όμως είναι ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται από ποιον, σε ποιον μεταδίδονται κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για την κυκλοφορία τα οποία στέλνουν τα αυτοκίνητα από μόνα τους. Είναι πάρα πολλά συστήματα ενσωματωμένα και αφορούν ε, την χρήση, την οδήγηση των οχημάτων. Ποια είναι λοιπόν τα δεδομένα αυτά, ποιος μπορεί να τα δει, τίθεται ζήτημα ιδιωτικής σφαίρας και προστασίας των δεδομένων. Λοιπόν, κόστος, κόστος στον ιδιωτικό τομέα και προστασία δεδομένων. Μάλιστα. Βιμ Φαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη σχετίζεται κάπως με αυτό το οποία είπε η κυρία Μάισνερ για τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει κάποια ανησυχία στους Ευρωπαίους για το ότι τα συστήματα αυτά της κυκλοφορίας μας παρακολουθούν. Δεν μου έρχεται τώρα και η Ολλανδική λέξη. Ε, και δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι επιθυμητό αυτό. Και μας είπε η κυρία εδώ πέρα πως δεν μπορούν να εξατομικευθούν τα δεδομένα ή να δούμε ότι αφορούν το συγκεκριμένο όχημα αλλά με βάλεσε σε η κυρία Μάισνερ. Και πώς θα αποφύγουμε το να μας παρακολουθεί λοιπόν ο μεγάλος ε, αδερφός. Να μην ε, είναι αυτό το κύριο θέμα της συζήτησης ε, των συστημάτων αυτών. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις τεχνικές εξελίξεις. Βλέπω σε διάφορες χώρες πως τα συστήματα αυτά ε, παίρνουν, ε, αποκτούν ε, διαστάσεις και υιοθετούνται όλο και περισσότερο. Το ερώτημα λοιπόν είναι θα προλάβουμε ή μέχρι να εκδοθεί η πράξη κατεξιοδότηση θα μας έχει ξεπεράσει η αγορά. Αυτή ήταν η δεύτερη μου ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Πράγματι αυτή ήταν ε, η συζήτηση που είχαμε κάνει και με τον Επίτροπο για το δικαίωμα στη λύθη. Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ. Πράγματι ετέθη το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Δεν θα το επαναλάβω. Εμένα θα με ενδιέφερε το εάν ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η κατάσταση τώρα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την θέληση εισαγωγής ε, ενός τέτοιου συστήματος να σας πενθυμίσω το τι γίνεται στην Γερμανία, τη συζήτηση για τα διόδια, την πιθανή εισαγωγή τους και νομίζω πως ε, ούτως ή άλλως ε, εγώ έχω ζητήσει από την Κομισιόν εδώ και καιρό ένα γενικό master plan για την κυκλοφορία στην Ευρώπη με όλα τα μέσα μεταφοράς. Οπότε θα ήθελα να γνωρίζω ποιες δυνατότητες βλέπει εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες, ε, ποια είναι η στάση των κρατών μελών για την πρότασή της. Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω παρόμοιες αμφιβολίες και προβληματισμό για ένα συναφές θέμα. Μια και οι εξελίξεις ε, καθοδηγούνται ουσιαστικά από την αγορά. Και σωστή και εύστοχη ήταν η παρατήρηση του κυρίου Βίμ Βαντερκάμπ και για το τεχνικό θέμα των προδιαγραφών αλλά και το θέμα του κόστους. Θα βελτιώσουμε την ποιότητα των πληροφοριών με μια καταξουσιοδότηση πράξη. Πολύ αμφιβάλλω. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχα μια αντίστοιχη εμπειρία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και δεν ήταν θετικά τα αποτελέσματα. Το κόστος λοιπόν, τεχνική ε, διάσταση και αν πραγματικά θα πιάσουν τόπο τα χρήματα. Ευχαριστώ. Μέια Κίλουν. Σας ευχαριστώ. Και εμένα με απασχολεί αυτό το θέμα της προστασίας των δεδομένων, ε, της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα, το θέμα της ασφάλειας προσωπικά δεδομένα και προσωπικοί λογαριασμοί με πληροφορίες μπορούν να περάσουν στο σύστημα ή από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, από όχημα σε όχημα. Επίσης, ε, τι γίνεται με τα συστήματα διοδίδων, διοδίων. Και εκεί είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα με τα δεδομένα. να ελέγχονται δηλαδή οι οδηγοί για το πόσο γρήγορα και πόσο άσχημα οδηγούν, αυτό φυσικά τους ενοχλεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε το θέμα με κάποιες εταιρείε που θέλουν να συμβάλλουν στο θέμα της ασφάλειας της οδικής. Ε, οι ασφαλιστικές εταιρείε, γιατί πληρώνουμε πολλά χρήματα στις ασφαλιστικές εταιρείε. Πώς θα βελτιώσουμε την ασφάλεια λοιπόν γενικώ στις οδικές μεταφορές, ιδιαίτερα στους νέους οδηγούς. Το θέμα της ασφάλειας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της προστασίας των δεδομένων. και οι δυνατότητες που έχουμε για να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ η Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση πολύ συχνά μιλούμε για την έλλειψη συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς, την πολυτροπικότητα. Θα εξασφαλιστεί βελτίωση στο θέμα αυτό και με ποιο τρόπο. Έχετε σχετικές πληροφορίες για το πώς η τελευταία πράξη κατεξοδότηση θα συμβάλλει και στη βελτίωση της διατροπικότητας. Ευχαριστώ. Φυσικά. Βλέπω ότι έχει αρκετές δυνατότητες σε αυτό το σύστημα και δυναμικό, αλλά όπως και η κυρία Μάισνερ και ο κύριος Βάντερκαμπ, και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς, ε, σε τι βαθμό θα έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, να μην δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα παρακολουθεί τα πάντα σαν το μεγάλο αδερφό. Δεν θέλω αυτό το σύστημα να επισέρχεται στην ιδιωτική σφαίρα των ε, ανθρώπων. Έχω δηλαδή αντίστοιχο προβληματισμό με αυτόν της κυρίας Μάισνερ και του κυρίου Βάντερ Κάμπ. Κύριος Κόχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η θέση ενισχύ ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται από τη λειτουργία του Γαλιλαίου ή αν όχι πώς θα συλλέγονται τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ντελή. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τα εθνικά σημεία πρόσβασης. Ε, στο 6.3 αναφέρεται πως υπάρχει δυνατότητα δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη να έχουν ένα κοινό σημείο πρόσβασης. Και εδώ πέρα ανησυχούμε για την προστασία των δεδομένων Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν εδώ πέρα για να έχουμε κοινά σημεία πρόσβασης που θα αφορούν δύο ή και περισσότερα κράτη-μέλη. Πώς ε, συμμορφώνεται αυτό το θέμα με την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ. Παύλ Ντέλετσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μάλλον έχασα την εισαγωγή, ε, εκτός αν το είπε ήδη η ομιλήτρια, κατά πόσον υπήρξε ανάλυση αντικτύπου. Από ό,τι κατάλαβα είμαστε πρώτων ε, διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων, δεν ξέρω αν έχει ήδη γίνει κάποια αξιολόγηση και αν ναι, ποιο ήταν το πόρισμά της, αν μπορείτε να μας πείτε. Και αν θα εξεταστεί επίσης από το Συμβούλιο αξιολόγησης των αξιολογήσεων αντικτύπου. Ε, γιατί νομίζω ότι αυτό γίνεται κάθε φορά που μας υποβάλλεται μια κατεξιόδηση πράξη. Πολλές οι ερωτήσεις. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση της ε, εκπροσώπου της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους όσους ε, υπέβαλαν ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω κάποια ομαδοποίηση. Θα ξεκινήσω από το βασικό σας προβληματισμό, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη καταξιδότηση πράξη δεν αφορά συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές ε, δεν αφορούν δεδομένα που συγκεντρώνονται από μεμονωμένα οχήματα στις οδικές μεταφορές. Πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρε ε, που περιλαμβάνονται στι υποδομέ. Σε μεγάλο βαθμό οι πληροφορίες αυτές ήδη υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Και θέλουμε με την κατεξουδότηση πράξη να εξασφαλίσουμε την παροχή των πληροφοριών αυτών με αρμονισμένο τρόπο σε παρόμοιο επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης επειδή μιλήσαμε για εναρμόνιση του μορφότυπου των δεδομένων, θέλουμε με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες να παρέχονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Όταν όμως μιλούμε για εναρμόνιση, δεν εννοούμε εναρμόνιση των πληροφοριών καθ' αυτών. Η κατεξιδότηση πράξη αφορά το πλαίσιο και το πώς θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες, όχι το περιεχόμενο αναφέρθηκα στο παράρτημα που περιλαμβάνει τα είδη των πληροφοριών που παρέχονται και τα είδη των δεδομένων που συλλέγονται. Το πιο αφιλεγόμενο ίσως σημείο θα αφορούσε την μεταφορά στους, στα οδικά, οδικούς άξονες. Έχουμε έργα οδικά, ε, συνθήκες ε, κυκλοφορίας, επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, όχι τα, τα πραγματικ, τις πραγματικές ταχύτητες. Σε καμία περίπτωση δεν συγκεντρώνουμε πληροφορίες που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, αφορούν συγκεκριμένο όχημα. Και επίσης, ε, όπως σας είπα, ήρθαμε σε επαφή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και είναι εξωσημείωτο ότι όποιες και είναι οι προδιαγραφές, ε, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του ITS, του εφιού Συστήματος Μεταφορών, όλες αυτές ε, υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Και θα γνωρίζετε και τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων που ενισχύει όλες αυτές τις αρχές και επίσης υπάρχει το θέμα της ανωνυμίας των δεδομένων ή το δικαίωμα της λύθης. Όλα αυτά τα σημεία περιχαρακώνονται και στη νέα πρόταση αυτό όμω τα είπα παρεμπιπτόντω, γιατί επαναλαμβάνω, η συγκεκριμένη κατεξοδότηση πράξη δεν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση. Οπότε το θέμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο να αποφεύγετε τέτοια παραβίαση καλύπτεται. Η κυρία Μάισνερ ρώτησε για το κόστος. Έχουμε κάνει ανάλυση κόστους-οφέλους της συγκεκριμένης κατεξουδότησης πράξης. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία για όλες τις κατεξουδότησες πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη ήδη υπάρχουν κάποια στοιχεία του συστήματος ε, πληροφοριών για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Βέβαια θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, ιδιαίτερα στι πληροφορίε που δίνονται μεταξύ διαφόρων χωρών άλλων. Πάντως, με το νέο μορφότυπο που προβλέπεται στη συγκεκριμένη κατεξοδότηση πράξη, θέλουμε μία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων και φυσικά και μέσω των διοικήσεων και εκεί ίσω δημιουργηθεί κάποιο συμπληρωματικό κόστος. Τα κράτη-μέλη βέβαια έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν πόσες επιπλέον πληροφορίες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες θα προσφέρουν. Πάντως, στις διαβουλεύσεις που είχαμε με τα κράτη-μέλη, μας είπαν ότι το ετήσιο κόστος ε, το Σημείου Πρόσβασης που θα δημιουργηθεί με την κατεξοδότηση πράξης θα κυμαίνεται μεταξύ 20 ε, ε, και 50 Αυτό καλύπτει το, το, την ε, κάλυψη, το επίπεδο περιπλοκότητας, το πώς θα δημιουργηθεί το σύστημα και πώς θα εφαρμοστεί. σε ό,τι αφορά τα εθνικά σημεία πρόσβασης και αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοση πληροφοριών μη επιτρεπόμενων, αν υπάρχει μια λύση που εφαρμόζει ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. Την πρόταση αυτή την περιλάβαμε στην κατεξοδότηση πράξη μετά από εκτενείς συζητήσεις που είχαμε με τα κράτη-μέλη. Και όπως είπα και στην αρχή, τα σημεία πρόσβασης θα καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές, ε, είτε αστικές, είτε υπεραστικές ε, επικοινωνίες ή συγκοινωνίες μεταξύ των πόλων και τα κράτη-μέλη μας ε, ζήτησαν τα σημεία πρόσβασης να καλύπτουν περισσότερα κράτη-μέλη για συγκεκριμένες διασυνοριακές περιοχές. Πάντως η ανταλλαγή πληροφοριών, όταν, είπα, όταν μίλησα για ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ πληροφορίες για την κατάσταση ε, των δρόμων, για την κατάσταση της κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη κατεξοδότηση πράξη δεν προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένα μεμονωμένα άτομα, συγκεκριμένα ταξίδια ή μεταφορά με συγκεκριμένα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Είχαμε επτά συνάντησεις όπως έλεγα με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ιδιαίτερο σε σχέση με την ε, εξοδότηση αυτή θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι όποια λύση δεν θα είναι κάτι που θα εξαναγκάσει τα κράτη-μέλη να πάνε σε απολύτως καινούργιες λύσεις. Ψάχνουμε τις διασυνδέσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί, που δεν υφίστανται για να βελτιώσουμε το σύνολο του συστήματος. Τα missing links. Σχετικά με την καθυστέρηση της εξιοδότησης αυτής, ρώτησε κάποιος, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, διότι αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον ίδιο τρόπο και δεν είναι διαθέσιμα στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτή η εξοδότηση θα επέτρεπε, εφόσον χρησιμοποιηθούν αυτές οι νέες υπηρεσίες, να υπάρχει ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας των δεδομένων αυτών, ώστε να υπάρχει μια εναρμονισμένη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η κυρία Κούλονεν ερώτησε σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και κατά πόσον τα δεδομένα για τα οποία μιλούμε μπορεί να προέρχονται από κόμβους επί του οχήματος επαναλαμβάνω ότι η εξοδότηση αυτή δεν εξετάζει τα λεγόμενα cooperative systems, όπου τα οχήματα είναι το κέντρο της όλης επικοινωνίας. Μιλούμε όμως για δεδομένα που κοιτούν την κυκλοφορία ως ενιαία οντότητα και όχι τα μεμονωμένα οχήματα. Επίσης για το intermodality που ρωτήσατε κυρία Ντέλη. Εδώ ψάχνουμε τις πληροφορίες, την ενημέρωση που έχουν σχέση με την κυκλοφορία. Όταν μιλούμε για το σχεδιασμό ενός ταξιδιού ή μιας μεταφοράς ή μεταφοράς προϊόντων για τις επιχειρήσεις, είναι τμήμα των διατροπικών ε, πληροφοριών, δεδομένων που αναζητούμε για τη βελτίωση του συνόλου των συστημάτων ε, ευρωπαϊκών μεταφορών. Και μιλούμε για το κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο ε, μεταφορών. Θεωρούμε ότι όταν αυτές οι πληροφορίες, αυτά τα δεδομένα στα σημεία πρόσβασης θα είναι διαθέσιμα, αυτό θα έχει πολύ σημαντική αξία και για τους διοργανωτές, διοργανωτές μεταφορών, είτε επιβατικών είτε μεταφορών προϊόντων, ώστε καλύτερα να σχεδιάζουν τη χρήση που θα κάνουν των υφισταμένων ε, συστημάτων μεταφοράς. Για τη σχέση μεταξύ αυτών των δεδομένων και των δυνητικών εξελίξεων στο ε, πλαίσιο του Γαλιλαίου, έχουμε πολλές πληροφορίες αυτή τη στιγμή με, τα, ε, με τις περαιτέρω εξελίξεις που μπορούμε να περιμένουμε των υπηρεσιών Γαλιλαίο μπορούμε να περιμένουμε πιο απτές εξελίξεις ή βελτιώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως τα δεδομένα αυτά δεν θα βασίζονται τόσο πολύ στα συστήματα ε, πλοήγησης ε, δορυφόρου αλλά θα στηρίζονται στα χερσαία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει συστήματα. Σχετικά με πληροφορίες που θα προέρχονται από δορυφορικά συστήματα, αυτά θα μπορούσαν να μας προσφέρουν περαιτέρω και καλύτερη κάλυψη του συστήματος στην Ευρώπη, και αναλόγως προς τις εξελίξεις της τεχνολογίας μπορούμε να προβλέψουμε διατάξεις αντιστοίχων προχωρημένων τέτοιων αν θέλετε συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών. Και για την τελευταία ερώτηση που σημείωσα, καθότι μιλούμε για κατεξιότητα πράξη, βεβαίως και κάναμε ανάλυση κόστους ωφέλους για τα συστήματα αυτά ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Διαβουλευθήκαμε τακτικότατα ιδιωτικούς φορείς ενδιαφερομένους, βεβαίως και εξωθείται από την αγορά και βεβαίως ε, οι ιδιωτικοί χρήστες, ε, υπηρεσίες, γραφεία που ασχολούνται με τις μεταφορές και τα ταξίδια, μας λένε συνεχώς ότι λείπουν πράγματα και ότι η ποιότητα των ε, δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκής. Ε, ευχαριστώ. Το τελευταίο λόγο έχει η κυρία Μάισνερ αν το θέλει. Ε, είμαι πολύ ικανοποιημένη από τις πληροφορίες αυτές. Νομίζω δεν έμεινε καμία ερώτηση αναπάντητη. Οπότε θα περιμένουμε την εξέλιξη της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στα διάφορα. Αν δεν υπάρχει και εδώ πέρα τίποτα, η επόμενη συνεδρία είναι Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Λύεται η συνεδρίαση, ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών.